Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε και σήμερα το πρωί, το δεύτερο ήμιση τη συνεδρίασής μας, έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε και να ψηφίσουμε. Έχετε τις κάρτες σας? Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω έτσι, εντάξει. Η πρώτη ψηφοφορία είναι η έκθεσή μας για ειδικά μέτρα για επιπλέον αρρωγή στις χώρες μέλη που επηρεάζονται από φυσικές καταστροφές. Έχουν ε, γίνει πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα για αυτά τα θέματα. Είχαμε τριμερή διάλογο για το Συμβούλιο. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα καταλήξαμε σε μια τελική λύση με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και μετά από όλα αυτά το πιο σημαντικό που θέλω να πω σε όλους εδώ είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους κοιόδης εισηγητές και προς τους συντονιστές επίσης των πολιτικών ομάδων για την στήριξή τους, την κατανόησή τους και την ε, τόσο έγκαιρη αντίδρασή τους, γιατί μόνο έτσι μπορέσαμε και να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε στο αίτημα του Συμβουλίου και να ολοκληρώσουμε την υπόθεση αυτή πριν από το καλοκαίρι. Συνεπώς ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους σας για τη στήριξή σας και την κατανόησή σας όσον αφορά την αξία της υπόθεσης αυτής. Λοιπόν, οι εισηγητές, αν θέλουν κάτι να πούνε, παρακαλώ, κύριος Βόγκαν. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι όλοι τα καταφέραμε πολύ καλά να καταλήξουμε σε συμβαστική συμφωνία. Και είναι πολύ σημαντικό που πέρασε στις πολιτικές ομάδες. Δεν ήταν εύκολο, το καταφέραμε στην Επιτροπή μας και μετά πήγαμε στον τριμερή διάλογο, όπως ξέρετε, με τους συναδέρφους και το Συμβούλιο ήταν πολύ απόλυτο δεν ήταν διατεθειμένο να βγει από το 90% της χρηματοδότησης. Τώρα Παρόλο που ήμασταν ε, απεσιόδοξοι, καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό, να αλλάξει τη θέση του και το Συμβούλιο. Τώρα έχουμε ένα συμβασμό που αποτελεί μια καλή συμφωνία. Είναι βέβαια συμβιβασμό. Όπω κάθε συμβιβασμό ε, σημαίνει ότι δεν ε, τα πετύχαμε όλα, αλλά νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτό. Ο κ. Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Δεν συζητάμε τις τεχνικές λεπτομέρειες, συζητάμε το σύστημα της πολιτικής συνοχής. Οπότε το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι να το αλλάξουμε ή να το καταστρέψουμε ή να το χρησιμοποιήσουμε για έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια πολύ ειδική μέθοδος για την Ιταλία. Δεν θελήσαμε βέβαια να αλλάξουμε ολόκληρο το σύστημα, Γι' αυτό και πιστεύω και εγώ ότι ο συμβασμός είναι καλός και καταφέραμε να έχουμε αυτό το όριο το οποίο τελικά σώζει το σύστημα. Δεν αλλάζουν όλα. Και αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, νομίζω. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Άλλος κανείς? Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε, και πάλι σας ευχαριστώ και να ψηφίσουμε τότε. Πρόκειται για μια ονομαστική ψηφοφορία, μια και μοναδική, ναι ή όχι. Συνεπώς, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Έχουμε ομοφωνία. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία που έχουμε για σήμερα, που είναι η έκθεση του κύριου Ομερζέ. Πρόθεση της συνοχής και της ανάπτυξης της εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμογή του άρθρου 349 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο Μερζέ, θέλετε κάτι να πείτε. Όχι. Καλώς. Συνεπώ, αρχίζουμε ευθύ αμέσω με την ψηφοφορία. Και αρχίζουμε με τη συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πιστεύω. Τώρα πάμε στη συμβαστική αριθμός 6. Ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην ε, τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 40. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται πράγματι. Τροπολογία 41. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει αυτή. Καταπίπτει, οπότε περνάμε στη συμβαστική 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 94 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 όχι, η άγκρη 12 καταπίπτει, οπότε πάμε στην 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρη 2. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 3 υπέρ κατά Α, ναι, σε δύο τμήματα έχετε δίκιο πάλι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 3. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 4, καταπίπτει και 5 και 6, φτάνουμε στην άγκρι 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 21, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 22, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 23, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Θέλετε να ελέγξουμε, ωραία. Άγκρι 23. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Λυπάμαι για το λάθος. Η 26 καταπίπτει και πάμε τώρα στη συμβαστική 17. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Άγκρι 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, να ελέγξουμε. Τροπολογία 106. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Λυπάμαι. Και πάλι να σηκώνετε τα χέρια σας, παρακαλώ. Πάμε τώρα στην συμβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 111 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 112. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 129. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε. 129. Τροπολογία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της φοφορίας. εγκρίθηκε. Συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η άγκρη 13 καλύπτεται από τη συμβαστική. Περνάμε τώρα στη συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά να ελέγξουμε καλύτερα για την Άγκρι 25 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. Κάποιο σχόλιο εκτός μικροφώνου, δεν ακούσαμε. 9 υπέρ, 15 κατά, λέει η πρόεδρος. Και μία αποχή, αν δεν απατώμε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ακολουθούμε, παρακολουθούμε την οθόνη όλοι για να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Τροπολογία τώρα 157 και 158 μαζί για την ίδια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 159. Με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης. Όχι, ωραία. Με την τροποποίηση αυτή. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω. Τώρα πάμε στην 186. 186. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 192. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 194. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197. Υπέρ, Αποσύρθηκε. Δεν το βλέπω στον καταλογό μου, αλλά εντάξει, καλώς. Συμβαστική 29 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 209. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 216. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 219. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 220 καταπίπτει, 221 τώρα. Όχι. Έχει εγκριθεί 220, πρέπει, 220 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα 221 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογίες 229, 230, Όχι, η 231 καταπίπτει, οπότε 229 και 230 μαζί υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 229 και 230. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτονται. ...232 έχει αποσυρθεί. 233 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 233. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Α, όχι, λυπάμαι, έχετε δίκιο. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 231 πρώτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα είπαμε 232 έχει αποσυρθεί και 233, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, καλά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, 233. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστικά 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 245 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 246 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 260 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 262 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 263 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ...270 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 271 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 274 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 275 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 276 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2,77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2,78 και 2,79 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 2,80 υπέρ έχει καταπέσει. 2,81 έχει καταπέσει. Περνάμε τώρα στην 2.82 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.84 απεσύρθη. 2.85 κατέπεσε. 2.86 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.087 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 288 υπέρ κατά αποχές δεκτή 289 υπέρ κατά αποχές δεκτή 290 υπέρ κατά αποχές δεκτή 291 υπέρ κατά αποχές δεκτή 292 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.93 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 ή μάλλον 14 υπέρ και 15 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 18 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Δεν ζητείται έλεγχος, οπότε και δεν τον κάνω. καλά, εντάξει, ας το ελέγξουμε. Την 22 λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Άγκρι B αγγλικό έχει καταπέσει. C, D, E, F, G καταπίπτουν όλα. Λοιπόν, τελική ψήφος, ηλεκτρονική κλίση ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή λοιπόν η έκθεση. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες για σήμερα στην Επιτροπή μας. Και τώρα ξέρετε ότι έχει αλλάξει το πρόγραμμά μας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αμαρτζή για να μας παρουσιάσει με λίγα λόγια τα αποτελέσματα της επίσκεψης στις Αζόρες της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο κύριο Μαρτζή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εδώ τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία και ε, για την στήριξή τους στις απότερες απόκεντρες περιοχές. Πράγματι πήγαμε στις Αζόρες για τρεις μέρες. Επιβεβαιώσαμε την συνέχιση της στήριξής μας στις απότερες απόκεντρες περιοχές. Εμείς κάναμε την αποστολή αυτή για να μπούμε στην ουσία αν θέλετε των προβλημάτων που φύγουν τις περιοχές αυτές και ίσως και το σύνολο των περιοχών που μας ενδιαφέρουν σήμερα. Η αποστολή μας λοιπόν ήταν κάτι το οποίο ε, προκάλεσε ενδιαφέρον από τις, το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών και η επίσκεψή μας αναφέρθηκε ευρύτερα και στον εθνικό τύπο και στον περιφερειακό τύπο της Πορτογαλίας. Λοιπόν, πριν περάσω στην ουσία, να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων για τη συμμετοχή τους και για την επικοδομητική τους συνεισφορά στην αποστολή στις Ασόρες. Όπως επίσης και για την φιλική ατμόσφαιρα και την ατμόσφαιρα την συνεκτική η οποία κυριάρχησε. Να ευχαριστήσω επίσης και το σύνολο του προσωπικού της Επιτροπής μας, τους τεχνικούς, την επιμελητία γενικά, οι οποίοι πήραν μέρος ε, στην ε, προσπάθεια αυτή. Τώρα για την ουσία γνωρίζετε ότι οι απότερες αυτές περιοχές υιοθέτησαν ένα μνημόνιο το οποίο ονομάζεται Μνημόνιο των Προέδρων των περιοχών αυτών, είναι αν θέλετε το πολιτικό έγγραφο, το οποίο αναδεικνύει τις βασικές διεκδικήσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αυτό το έγγραφο κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν από την επεξεργασία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια στρατηγική για τις απόκεντρες περιοχές. Και ε, το έγγραφο αυτό κυκλοφόρησε τη στιγμή που η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή υιοθέτησε την έκθεσή της για την εφαρμογή του 149, το οποίο άλλωστε υποστηρίξατε σήμερα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κομβική στιγμή για τις απόκεντρες περιοχές και η αποστολή μας ε, έτυχε να πάει σε μια σημαντική συγκυρία και πράγματι οι αρχές ε, των Αζόρων περίμεναν από μας να εκφράσουμε τις θέσεις και τα προβλήματα τα οποία ε, μας ε, χαρακτηρίζουν τα εγγραφά μας. Στις ασόρες ειδικότερα δίδεται μεγάλο βάρος στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Η πρώτη συνάντηση, δεν χρειάζεται να ιεραρχήσω τις συναντήσεις γιατί ήταν όλες ενδιαφέρουσες, και σημαντικές, αλλά η βασική συνάντηση την οποία είχαμε ήταν με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Κυβέρνησης και ακριβώς είχε αυτό το θέμα. Η αντιπροσωπεία μας συγκράτησε από τον πρόεδρο των Αζωρών δύο βασικά μηνύματα. Πρώτον, και προφανώς οι Αζόρες ανησυχούν. Ανησυχούν για την διατήρηση μιας πραγματικής περιφερειακής πολιτικής προστασίας η οποία βασίζεται, εδράζεται, αγκυρώνεται πάντα στις αρχές της αλληλεγγύης απέναντι στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα τις απόκεντρες περιοχές. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο είναι πιο συγκεκριμένο και αυτό ακούστηκε δυνατά στις Αζόρες κίνδυνος εκφυλισμού της πολιτικής αυτής μέσω του πολλαπλασιασμού των χρηματοδοτικών μέσων. Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης επανειλημμένα μας είπε ότι είχε αυτήν την ανησυχία και όταν τον συνάντησα σε προσωπικό επίπεδο μου είπε ότι περίμενε από την Επιτροπή μας να δώσουμε μάχη στα πλαίσια του προγραμματισμού για μετά το 2020 έτσι ώστε να διατηρηθεί για τις περιφέρειες αυτές το καθεστώς των επιδοτήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αζόρες ε, είναι χρικές στα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά τα μέσα είναι λιγότερο ελκυστικά για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές που είναι απομεμακρυσμένες από την υπηρετική Ευρώπη και όχι τόσο για τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο, αν θέλετε, των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα. Μετά επισκεφθήκαμε, κάναμε κάποιες επισκέψεις μάλλον, που μας επέτρεψαν να επιβεβαιώσουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια καταναλώνονται ορθά ε, στις απότερες αυτές απομεμακρυσμένες περιοχές και ότι Ακριβώς όπως είχαμε πει στα τελευταίες συναντήσεις μας, ε, έχει υπάρξει μια θεματολογική συγκέντρωση των πιστώσεων ε, με στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Έτσι λοιπόν εμείς ε, πολλαπλασιάσαμε τις παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχει μια πραγματική δυναμική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των περιοχών αυτών. Και αυτό το οποίο είπα είναι ότι αναφερόμεθα στις απότερες αυτές περιοχές υπό το πρίσμα ε, του προβλήματος, του χάντικαπ το οποίο παρουσιάζουν, του μειονεκτήματος, λόγω του απομεμακρυσμένου χαρακτήρα τους. Αυτό το οποίο λέγω επίσης είναι ότι η γεωγραφία για τις Ασόρες είναι και το βασικό του πλεονέκτημα, διότι ακριβώς η γεωγραφική της θέση καθιστά τις Αζόρες κέντρο του Ατλαντικού, σε ένα γεωστρατηγικό σημείο σημαντικό, ένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα, το οποίο μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι στις αζόρες πολλά πράγματα είναι αυτά τα οποία εξελίσσονται ε, με σωστό τρόπο. Η γεωγραφία έχει δώσει την δυνατότητα για μια τρομακτική βιοπικιλότητα είναι μια ηφαιστειογενής χώρα η οποία θα έλεγα τροφοδοτεί τις ανάγκες της ενέργεια από τη γεωθερμία και μπορεί να διεκδικήσει την ενεργειακή αυτονομία. Η γεωγραφία και ο νησιωτικός χαρακτήρας δίδει την δυνατότητα αξιοποίησης της θαλάσσιας οικονομίας, της κιανής οικονομίας και γι' αυτό ακριβώς είδαμε με συγκεκριμένο τρόπο το τι γίνεται στις περιφέρειες αυτές, έτσι ώστε οι Αζόρες να μπορέσουν να ηγηθούν σε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, ε, προς όφελός τους βέβαια, αλλά και προς όφελος όλων των γαλλικών και ευρωπαϊκών απότερων μεμακρυσμένων περιοχών. Η γεωθερμία, η φεστιολογία, Υπάρχει ένα κέντρο βέλτιστων πρακτικών πανεπιστημιακό στον τομέα της ηφαιστειολογίας και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα και με τα πανεπιστήμια των αντιλών της Καραϊβικής γενικότερα. Έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός πλεονεκτικού για όλους τρόπους συνεργασίας. Αυτά λοιπόν. Όταν μετακινούμεθα στις περιφέρειες αυτές, νομίζω ότι καλό θα ήταν στο πρόγραμμα να προβλέπουμε ε, την εξέταση των βασικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές. Διότι οι δείκτες και οι αριθμοί τους οποίους ε, έχουμε αποδεικνύουν κάποια ποσοστά ανεργίας υψηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, μας δείχνουν επίπεδα ένδυας υψηλότατα επίσης, δηλαδή ανάβουν κόκκινα φωτάκια σε πάρα, πολλές, ε, ε, σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι λοιπόν σωστό από τη μία να διαπιστώνει κανείς ότι το λειτουργικά προγράμματα εφαρμόζονται με συγκεκριμένους και συμβατούς στόχους, που μπορούν να επιτρέψουν να πετύχουμε τους αρχικούς ε, στόχους, από την άλλη όμως ε, δεν πρέπει να αγνοούμε το μέγεθος των δυσκολιών, γιατί οι αποστολές αυτές μερικές φορές θα έλεγα ε, στρεβλώνουν την τελική εικόνα, γιατί γίνεται μια προσπάθεια και από τους τοπικούς παράγοντες να δείξουν ότι όλα γίνονται όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεχνούν να μας δείξουν ποια είναι τα δύσκολα τα οποία αντιμετωπίζουν. Αλλά είμαι βέβαιος ότι οι περισσότερες από τις αντιπροσωπείες σε αυτές τις χώρες βλέπουν ποιες είναι οι δυσκολίες Βλέπουμε τι γίνεται με την εξαφάνιση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που στις Αζόρες όπως και στη Μαδέρα δημιουργούν επιπλέον προβλήματα τα οποία και η δική μας Επιτροπή πρέπει να ερευνήσει έτσι ώστε να κάνει κάποιες αντισταθμιστικές προτάσεις στην Επιτροπή Γεωργίας. Λοιπόν, γενικά η αποστολή ήταν ενδιαφέρουσα, νομίζω και παραγωγική και είμαι βέβαιος ότι θα εντάξουμε από εδώ και πέρα στη συνέχεια των εργασιών μας αυτά τα οποία είδαμε και μάθαμε στις Αζόρες. Ευχαριστώ. Ε, α, έχετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Μου δίνετε το λόγο θα ήθελα να πω ξεκινώντας... Ε, θα ήθελα να πω ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι απότερες αυτές περιοχές είναι διαφροτικού τύπου και το βασικότερο των προβλημάτων είναι οι μεταφορές. Ε, γιατί η Μαδέρα επίσης είναι δύσκολη κατάσταση και σε επίπεδο κόστους Υπάρχουν ε, επιπλέον διαρθρωτικές επιπτώσεις από τις δυσκολίες της μεταφορές και η οικονομία η τοπική δεν μπορεί εύκολα να είναι ανταγωνιστική. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επηρεάσει τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ με τους δύο προηγουμένους συναδέλφους. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη, τη γραμματεία της ομάδας. Θα προσθέσω και δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν εξεπλάγει ευχάριστα βλέποντας ότι οι Αζόρες όπως και όλες οι εξόχως από κεντρές περιφέρειες δεν είναι μεν σε ε, θετική θέση, αλλά την ε, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση την αντιμετώπισαν πολύ καλά, καλύτερα από άλλες περιοχές, ακόμα και στην ίδια την Πορτογαλία. Πρόκειται για μια επιτυχία των Αζωρών και τα διαρθρωτικά ταμεία σίγουρα συνέβαλαν και αυτά στο καλό αποτέλεσμα. Δεύτερον, στις Αζόρες ε, επισκεφθήκαμε δύο νησιά. Αλλά βλέπουμε παντού τη γαλάζια σημαία με τα χρυσά αστέρια. Αυτό έχει αξιοποιηθεί και πρέπει να το αναδείξουμε. Πάρα πολλά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, βοηθούν την ανάπτυξη των αζωρών. Αυτό που με ενόχλησε λίγο ήταν ότι η σχετική επικοινωνία πολλές φορές δεν είναι τόσο επιτυχής όσο θα φανταζόμαστε. Για παράδειγμα, πήγαμε σε ένα νηπιαγωγείο, βρεφονηπιακό σταθμό, εξαιρετικό, πολύ θα ήθελαν ε, με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ε, δεν γνώριζαν εκεί πόσα χρήματα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο αυτό και είναι κρίμα, γιατί ένα τέτοιο έργο σε μια ε, οικιστική περιοχή που μπορεί να αξιοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους, είναι κρίμα να μην γνωρίζουν το ιστορικό και τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριλάβουμε στις διαπιστώσεις μας και αυτό το θέμα, ότι δηλαδή θα πρέπει να κοινοποιούνται τα έργα καλύτερα. Επίσης επισκεφθήκαμε ένα κέντρο τεχνολογίας και αυτό επίσης ενόχλησε λίγο γιατί η κυρία που έκανε την παρουσίαση είπε πολλά πράγματα αλλά όταν έγιναν ερωτήσεις μας είπε ότι δημιουργήθηκαν μόνο τέσσερις θέσεις εργασίας. Πράγμα παράδοξο. Και εκ των υστέρων απεδείχθη ότι δεν ήταν σωστό. Ίσως δεν έγινε κατανοητή η ερώτηση. Στην επιχείρηση που διαχειρίζεται το κέντρο τεχνολογίας δημιουργήθηκαν τέσσερις θέσεις εργασίας, αλλά δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα ήταν πόσοι εγκαταστάθηκαν εκεί στο κέντρο καινοτομίας και πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν εκεί. Αυτό διευκρινίστηκε σε μετέπειτα ε, ερωταπαντήσεις. Ε, σε μια επιχείρηση, σε μια επιχείρηση ε, μάθαμε αργότερα ότι δημιουργήθηκαν 50 θέσεις εργασίας αφού η επιχείρηση εγκαταστάθηκε εκεί. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνιακή. Και στο τέλος, ε, όταν μιλήσαμε με τους εκπροσώπους του Δημάρχου, ε, είδα ότι έγινε αθέμητη κριτική στην Ευρώπη, ότι δηλαδή το ένα δεν πάει καλά, το άλλο δεν λειτουργεί, πρόβλημα με την κατασκευή δρόμων, ε, ότι έμπλεξαν αποφάσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης. Δηλαδή υπήρχαν κάποια θέματα. Όταν δηλαδή κάποιος διαθέτει και χρησιμοποιεί πολύ ικανοποιητικά κάποια κονδύλια σε μια τέτοια εξόχως από κέντρη περιφέρεια, ε, νομίζω ότι καλό θα ήταν να προβληθεί επικοινωνιακά το έργο αυτό, να γίνει κατανοητό δηλαδή από τον κόσμο πραγματικά ότι όντως υπάρχει μια μεγάλη προθυμία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, να καταδειχθεί η ελληνική και αυτό γίνεται έμπρακτα. Ο κύριος Ομαρζέ ε, και άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για πολλά θετικά, ε, αλλά όλα αυτά με έκαναν να σκεφτώ ότι το μήνυμα, τα αποτελέσματα, τα καλά θα πρέπει να περάσουν και στον κόσμο εκεί. Ευχαριστώ. Κύριο Βον, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρζέ για το πώς προείδρευσε στην αντιπροσωπεία που ήταν εξαιρετική. Ε, όπως πάντα είχαμε πάρα πολλή δουλειά, δεν προλάβαμε να δούμε λίγο την τοπική κουλτούρα. Λίγο το βράδυ. Ε, Τρία πράγματα μου κάνανε εντύπωση από την επίσκεψη. Κάποια κονδύλια χρηματοδοτούν κάποιες βασικές υποδομές σε ένα σχολείο, πήγαμε σε ένα σχολείο, αλλά ε, υπήρχαν και οικονομικά έργα. Ε, πήγαμε σε ένα λιμάνι, σε ένα κέντρο πάρκο καινοτομίας, ε, αλλά ορισμένα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση ήταν ότι αυτή τη στιγμή ε, οι προβλέψεις στηρίζονται όχι τόσο στο αποτελέσματα όσο στις εισρωές εκροές. Στις Αζόρες και σε άλλες ε, απόκεντρες περιοχές ε, θα πρέπει στον επόμενο γύρο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στις, στην απόδοση. Θα πρέπει να δείξουμε δηλαδή τις δυνατότητες εκπαίδευσης που θα δώσουν απασχόληση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει και γρήγορα. Επίσης μου έκανε εντύπωση το ποσοστό συγχρηματοδότησης κάποιων έργων που ήταν περίπου 85% σε πολλά έργα που επισκεφθήκαμε. Ίσως και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Ε, μπορεί δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πιο βιώσιμα τα έργα αυτά. Τέλος, ε, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στα άλλα έργα μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί δικαιούχοι είτε δεν εγνώριζαν τον αντίκτυπο των ενωσιακών κονδυλίων και σίγουρα δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες, δηλαδή πόσο συνέβαλαν τα κονδύλια στα έργα στα οποία ε, απασχολούνταν. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, όχι μόνο σε σχέση με τις Αζόρες, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε πέρσι τον Ιούνιο το δημοψήφισμα για τον Brexit και σε πάρα πολλά έργα και εκεί πολλοί δικαιούχοι δεν γνώριζαν ε, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και εκείνοι που εργάζονταν στα έργα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ε, δείξουμε στον κόσμο τι χρηματοδοτεί και τι κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Μαλέτριτς. Και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον κύριο Μαρζέ που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας. Ήταν εξαιρετική εμπειρία που είδαμε επιτόπου τα έργα αυτά. Σημερίζομαι και την αίσθηση αυτή που ανέφεραν οι συνάδελφοι σε σχέση με τους στόχους και τι πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους. Όπου και να ρωτήσαμε για τους στόχους και τι ήθελαν να επιτύχουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεν πήραμε απαντήσεις ιδιαίτερα στη βιβλιοθήκη, γιατί είναι ένα τεράστιο κτίριο αυτό στο μέσο ενός μικρού νησιού και δεν ήξεραν να μας εξηγήσουν τι έπρεπε να κάνουν με αυτό το κτίριο, πώς να το χρησιμοποιήσουν και πώς να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάπτυξη μέσω αυτού στο νησί. Εξεπλάγιν θετικά όταν συζητήσαμε με τον πρόεδρο, ο οποίος μας εξήγησε ότι πάντα είχαν οικονομική ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια, γύρω στο 10-11% που είναι πάρα πολύ ψηλό ε, ποσοστό ανάπτυξης και είπε ότι δεν είχαν προβλήματα με την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα γιατί αυτά που επενδύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τους βοηθούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Σε στρατηγικό επίπεδο συζητήσαμε μαζί του όλα τα ζητήματα αυτά που μας απασχολούν και εδώ για την πολιτική συνοχή και συμφώνησε λέγοντας ότι παρόλο που δεν έχει με μακροοικονομικές ερεσιμότητες προβλήματα, όμως συμμερίζεται την άποψή μας ότι δεν είναι σωστό να συνδέουμε την πολιτική συνοχής με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε. Τα συζητήσαμε αυτά σε σχέση με το μέλλον, γιατί θέλαμε να ακούσουμε από την πρακτική τους εμπειρία τι πιστεύουν για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και εκείνοι είπαν ότι θέλουν παρόμοιους κανόνες, αλλά και αλλαγές σχετικά με αυτή τη σύνδεση που γίνεται με την οικονομική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε Βαν Νίστελ Ρόι. Εγώ δεν ήμουν στην αντιπροσωπεία. Α, θα, θα μιλήσω αργότερα. Και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρζέ, ο οποίος ε, προείδρευσε εξαιρετικά. Συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις που ακούσαμε είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εργαστούμε για την ορατότητα. Για την τελευταία παρατήρηση είναι μια ε, γνώμη αυτή. Αυτή είναι η γνώμη ενός Προέδρου της Ένωσης των Κοινοτήτων, ο οποίος είπε ότι θέλει τα κονδύλια να επενδύονται σε δρόμους. Αυτό είναι η επιθυμία του ενδεχομένως, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς στα πλαίσια ενός πλαισίου πολιτικής για το 2020. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο θεματικά, εξεπλάγιν διότι ε, χρηματοδοτούμε βασικές υποδομές, αλλά αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών να ε, μεταφέρουν όλα αυτά στις περιφέρειες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούμε, για παράδειγμα, ένα νηπιαγωγείο, αυτό είναι βασική αρμοδιότητα των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων, όχι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν θα συνδέεται ε, προς την επιτυχία της στρατηγικής 2020. Ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που λέει ο κόσμος εκεί. Είναι δική μας ευθύνη και καθήκον να θέσουμε το πλαίσιο πολιτικής μετά το 2020 όμως. Και αυτό, όχι μόνο, αυτό δεν περιορίζεται στην έκφραση επιθυμιών ε, από την πλευρά του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι μόλις εκφράσουμε μια επιθυμία μέσα θα πρέπει να σπεύσουμε να ανταποκριθούμε πάντοτε. Ο κύριος Βανίστελ Ροϊ, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σόφρον να κάνουμε τέτοιες επισκέψεις σε αυτές τις περιοχές. Τώρα μια γενική παρατήρηση. Όταν κάνουμε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να τους επιτρέπουμε να βλέπουν ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή, δεν θέλουμε μόνο να τους δώσουμε μία ε, υποδομή, αλλά να τους εντάξουμε στη διαρθρωτική πολιτική. Να καταλάβουν τους στόχους σε έναν ορίζοντα πολλές φορές και δέκα ετών. Και νομίζω ότι αυτό λείπει. Γιατί θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε βάθος το τι κάνουμε και τι σημαίνει η πολιτική μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα πετύχουμε να έχουμε και συμμάχους επιτόπου με τους οποίους θα συζητούμε, θα κρίνουμε την πρόοδό τους και θα δούμε τι θέση είχε η πολιτική μας. Τον Ιούνιο θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια κοινή συζήτηση, να συζητήσουμε για την έκθεση Μπούντα γενικότερα, για την ορατότητα, για το τι κάνουμε και να προσθέσω ότι στο ΕΛΚ ε, ετοιμάσαμε ένα δημοσίευμα που θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο στην Ακροάση που λέγεται ε, «Ας αφήσουμε τα αστέρια να λάμψουν». Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει το έργο να τελειώνει όταν πληρωθεί και ο τελευταίος λογαριασμός. Θα πρέπει σε πολλαπλά επίπεδα να ε, γίνει η επικοινωνία ούτε θα πρέπει να κατηγορήσουμε τα κράτη-μέλη. Ε, ούτε θα πρέπει να αλληλό κατηγορούμεθα γιατί δεν κατασκευάστηκαν κάποιοι οδοί. Θα πρέπει να αναλυφθούν κοινέ δράσεις. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πάντως υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσης, θα υπάρξει και σχέδιο δράσης από την Κομισιόν και έτσι θα πρέπει να δουλέψουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και στο κοινωνικό ταμείο για την εκπαίδευση κλπ. Ε, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα έργα λοιπόν. Καλό ήταν που συζητήσαμε όλα αυτά. Το επόμενο σημείο θα είναι και το καινούριο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε εκεί θα ξαναέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Θα θα επανέλθουμε στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή, για την έκθεσή σας κύριε Ομαρσέ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πόσο ε, διαφορετική είναι η πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Για μας, στην Επιτροπή μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προέρχονται, να, να αποκομίζουμε εντυπώσεις από διαφορετικές περιφέρειες της Ευρώπης και το πώς λειτουργεί η πολιτική συνοχή ε, στις αυτές. Αυτό θα είναι χρήσιμο και για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις και αποφάσεις στην Επιτροπή Ρέτζη. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως με εντυπωσιάσατε γιατί μέσα σε δύο μέρες μόνο επισκεφθήκατε δύο νησιά, πάρα πολλά ε, μέρη, πάρα πολλά έργα. Πραγματικά είναι απίστευτο πώς το καταφέρατε. Ήταν πολύ επιτυχής η αποστολή αυτή και τα πήγε πάρα πολύ καλά η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ρέντζε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την γνωμοδότηση που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή Προπολογισμών. Η έκθεση είναι προετοιμάζοντας θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ε, πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2020. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων σήμερα λοιπόν για την γνωμοδότησή μας με τον κύριο Βόγκαν που είναι και ο εισηγητής μας για την γνωμοδότηση αυτή. Κύριε Βόγαν, παρακαλώ να υποβάλλετε έκερα την γνωμοδότησή σας πριν την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, που είναι στις 20 Ιουνίου, σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, οπότε έχετε και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ είναι πολύ σημαντικέ για όλου μα οι επόμενε πολιτικές δημοσιονομικέ προοπτικές. Χρειαζόμαστε τον κατάλληλο προπολογισμό για τι πολιτικέ μα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν μια καλή ιδέα να έχουμε πριν καθίσω και γράψω κάποιο κείμενο, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για να ακούσω τις απόψεις των συνοδέλφων για τα διάφορα ζητήματα. Πολλά είναι που πρέπει να συζητηθούν εδώ στην περιφερειακή πολιτική και μετά θα προσπαθήσω να τα βάλω και στο χαρτί και να έχω έτοιμο κάτι, όπως είπατε, στην επόμενη συνεδρίασή μας. Ποια είναι λοιπόν τα θέματα για τα οποία θέλω τη γνώμη των συναδέρφων. Το πρώτο είναι το μέγεθος του προπολογισμού. Όπως πάντα γίνεται στις συζητήσεις για τα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχει ο καυγάς δυστυχώς ανάμεσα στους καθαρούς εισφορείς και τους καθαρούς δικαιώχους. Αυτή τη φορά βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι στο τραπέζι όπως πάντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω από 10% δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Άρα τι θα γίνει, θα είναι πιο μικρός ο προπολογισμό, θα το δεχτούμε αυτό ή θα θελήσουμε να διατηρήσουμε τον προπολογισμό όπως έχει ή να τον αυξήσουμε και όλα. Και τότε ποιος θα βάλει αυτά τα λεφτά που θα λείψουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ψάξουμε να βρούμε νέα ε, δημοσιονομικά συστήματα χρηματοδότησης του προπολογισμού μας. Σίγουρα το συζητάει αυτό εδώ και καιρό η Επιτροπή Προπολογισμών. Τι θα γίνει με του ίδιου πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπω πρέπει αυτοί να αυξηθούν αντί να συζητήσουμε περισσότερα χρήματα από τι χώρε μέλη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θα είναι τι θα πάει από τα χρήματα αυτά στην περιφερειακή πολιτική. Την τελευταία φορά υπήρξαν σημαντικές περικοπές. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε, να αγωνιστούμε, να δώσουμε τη μάχη μας για την περιφερειακή πολιτική στον προπολογισμό. Κάποιοι στην Επιτροπή και όχι μόνο θέλουν περικοπές στην περιφερειακή πολιτική. Ε, κάποιες χώρες θέλουν ένα εντελώ νέο σύστημα. Να βασιστούμε περισσότερο σε δάνεια και όχι σε επιχορηγήσει. Συνεπώς πρέπει να δώσουμε τη μάχη μα για την περιφερειακή πολιτική στα πλαίσια του νέου προπολογισμού. Να δούμε επίση και τη νέα περίοδο πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Θα είναι πάντα εφταετής η περίοδο αυτή, όπω είδα και κατά το παρελθόν. Αυτό βολεύει την πολιτική συνοχή, αλλά από την άλλη μεριά δεν συμπίπτει με τι θητείε του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κάτι άλλο. Κάποιοι είπαν να είναι 5 συν 5 χρόνια. Είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε για την επόμενη περίοδο. Κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε είναι το πόση ευελιξία θέλουμε στην επόμενη περίοδο πολιετούς δημοσιονομικής προοπτικής. Χρειαζόμαστε ευελιξία στον προπολογισμό βέβαια για να κυκλοφορεί το χρήμα αν κάπου υπάρχει ε, υπο δεν έχουν ε, απορροφηθεί δηλαδή κονδύλια, μήπως μπορούμε να τα βάλουμε κάπου αλλού στην περιφερειακή πολιτική είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε με τα λίγα χρήματα που έχουμε. Τεχνική αρρωγή. Λοιπόν, καλή είναι η ευελιξία, αλλά πρέπει να βρούμε πώς αυτή η ευελιξία θα υπάρχει μεν, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα την παίρνουν, θα παίρνουν τα χρήματα από την περιφερειακή πολιτική για να καλυφθούν άλλες ανάγκες. Και τι θα γίνει με την μία απορρόφηση κονδυλίων. Εφόσον δεν δαπανώνται τα χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, τι θα γίνεται. Τα χρήματα πρέπει να παραμένουν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Γιατί να πηγαίνουν πίσω στις χώρες μέλη, θα μπορούσαν να δαπανηθούν στην περιφερειακή πολιτική, για παράδειγμα. Οπότε και αυτό πρέπει να το δούμε στη συζήτηση αυτή για τι επόμενε πολιτικέ δημοσιονομικέ προοπτικές. Πολιτική συνοχής. Τώρα, απλοποίηση. Πάντα μιλάμε για απλοποίηση, αλλά δεν έχουμε συζητήσει πραγματικά για το πώς θα απλοποιήσουμε και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την πολιτική συνοχής. Μιλάμε για το 1 συν 1, 2, 3. Κάποιοι, και συστήσαμε και με το ελεκτικό συνέδριο, δεν τους αρέσει. Θέλουν νη συν Τίποτα άλλο. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να πάμε πίσω στο νησιν 2. Άλλοι δεν θα το θέλουν. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε τι προτιμάμε εμείς. Άρα να το σκεφτούν οι συναδελφοί Και διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή. Εγώ όμως θα αρκεστώ σε αυτά. Ήθελα λοιπόν να σας τα θέσω αυτά, ώστε να τα σκεφτείτε και να σας πω ότι τέτοια ζητήματα θα θέλω να συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου του Ιουνίου. Υπάρχουν βέβαια και άλλα για τα οποία δεν μίλησα σήμερα. Θα τα συμπεριλάβω στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σκιώδης εισηγητές, παρακαλώ. Ποιος? Παρακαλώ, κυρία Τόμασιτς. Θέλετε Πρώτα κύριος Φανίστεροι. Ο κύριος Φανίστεροι. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε τις νέες πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ας ελπίσουμε ότι θα μας έρθουν όπως προβλέπετε, όπως έχουν σχεδιαστεί. Γιατί πρώτα είναι αυτό και μετά είναι το πρόγραμμα συνοχής. Η έκθεση συνοχής είναι για τα τέλη της χρονιάς μετά τι πολιτικές δημοσιονομικέ προοπτικέ. Συνεπώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να πιεστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να προχωρήσει. Γιατί αλλιώ πιέζονται όλα για το 2018 και 2019 που θα έχουμε και τις εκλογές και το Brexit. Όπω είπατε δεν διευκολύνει τα πράγματα το Brexit, μάλλον τα δυσκολεύει. Γιατί τι θα γίνει οικονομικά. Οπότε στο δεύτερο ήμιση της περίοδου αυτής είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ταχύτητα. Αυτό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταχύτητα για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Γιατί όσο περισσότερο περιμένετε, τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Δεύτερον, έχουμε την έκθεση για το ποια είναι τα θεμέλια μας, πού βασιζόμαστε, ποια είναι τα, τα βασικά. Πρέπει να μιλήσουμε για τη συνοχή αυτή καθεαυτή σε αυτό το στάδιο εξέλιξης της Ευρώπης. Γιατί βλέπουμε ότι η ολοκλήρωση βοηθιέται βέβαια από τη συνοχή για περιφέρειες και χώρες με τεράστια αποτελέσματα. Αν δείτε την περίοδο μετά τον κομμουνισμό τι έγινε στις διάφορες χώρες, πώς κυκλοφορεί η γνώση, πώς ε, στηρίζονται οι χώρες αυτές για το πώς να οργανωθούν καλύτερα και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης. Συνεργασία, πώς γίνεται στα διάφορα επίπεδα με τους διάφορους ε, εταίρους Και βέβαια έχει να κάνει αυτό και με τις ίδιες τις αρχές της συνθήκης. Η συνοχή είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Συνεπώς, να απορρίψετε συγχρόνως την ιδέα των ε, τριών ταχυτήτων. Ότι ο νικητής τα παίρνει όλα. Έτσι, αυτή είναι μία ταχύτητα, δηλαδή πια οι μεγάλες ε, πόλεις, μητροπόλεις στην Ευρώπη και κάποια άλλη κάτι λιγότερα και τα υπόλοιπα τα παίρνουν όλοι οι Κινέζοι. Το λιμάνι του Πειραιά, για παράδειγμα, αυτή είναι η Ευρώπη. Όχι. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που συζητάμε εμείς εδώ. Οπότε, όσον αφορά τις αναλλακτικέ, όσον αφορά την βασική κίνηση πίσω από την συνοχή, η συνοχή πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και από εκεί αντικατοπτρίζεται και ε, ο τρόπος με τον οποίο θα δούμε ε, τη νέα περίοδο πολιωτών προοπτικών, η οποία βέβαια χωρίζεται σε νέες προτεραιότητες, τη εξωτερικά σύνορα, μετανάστευση, ασφάλεια, ε, απασχόληση κλπ. Ναι, μέχρι τώρα όμως είχαμε και το δικό μας το τομέα, με πολλούς στόχους οι οποίοι στηρίζονται από την πολιτική συνοχής. Και εδώ είναι που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή. Τώρα είμαστε στη μέση της προηγούμενης περίοδου. Αν κάποιος ζητάει αποτελέσματα, η δικιά μας Επιτροπή έχει αποτελέσματα να επιδείξει. Και με κάποιες άλλες, περιβάλλον, εκπαίδευση και πολιτισμός. Οπότε δεν είναι τεχνικό το ζήτημα, είναι θέμα αρχών. Και η τρίτη μου παρατήρηση, κοιτάω βέβαια τη δικιά μου κατάσταση στην Ολλανδία πώς έχουν τα πράγματα. Η κυβέρνησή μου δεν στηρίζει ιδιαίτερα τη συνοχή. ως αυτό σκοπό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά μέσα και μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί όπως η μεγαλύτερη ειδίκευση, η χρήση της γνώσης σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, στην Γεωργία. Χτες συζητήσαμε, για παράδειγμα, για τα βιοπροϊόντα στη Γεωργία. Οπότε, ε, αφήνοντας τη γνώση να κυκλοφορήσει και χρησιμοποιώντας τα χρήματα, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και είναι η λογική απάντηση σε αυτό που λέμε the winner takes it all, ότι ο νικητής κερδίζει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να δουλέψουμε ε, με την πληροφορική για την βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται καλή σχέση λοιπόν ανάμεσα στην έρευνα και την ανάπτυξη στα πλαίσια του 2020 και να υπάρχει περιφερειακή εδαφική συνεργασία σε αυτό έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι θα υπάρχει περισσότερη στήριξη από ό,τι νομίζουμε όταν συζητάμε για την περιφερειακή συνεργασία. Κάτι το οποίο κάνει κάπως λιγότερο σκληρή την ε, πραγματικότητα. Η εξειδίκευση πιστεύω ότι στο μέλλον θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα πολύ συγκεκριμένα. Αυτή τη βδομάδα στο Ελσίνκι λαμβάνει η χώρα μια τεράστια διάσκεψη. Συμμετέχει και η Επιτροπή και πρόκειται ακριβώς για την ευφύ εξειδίκευση, για τις έξυπνες περιφέρειες, για το τι κάνουν ώστε να είναι προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Και από εκεί θα πετύχει η πολιτική μας, η περιφερειακή, Πώ θα πετύχει, προσφέροντας κονδύλια τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανείς όπως να είναι ή θέτοντας ε, μεγαλύτερους στόχους. Λοιπόν, επιτάχυνση. Αυτό χρειάζεται. Ευχαριστώ κυρία Τόμασιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική τα τελευταία χρόνια έγινε η βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και μέσον για την επίτευξη των μεγάλων πολιτικών στόχων μας και με τους συγκεκριμένους στόχους που προβλέπονται στις συνθήκες. Η πολιτική συνοχή θα συνεχίσει έτσι και μετά το 2020 και θα παραμείνει, πρέπει να παραμείνει, πολιτική συνοχής για όλα τα κράτη-μέλη. Η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να αποδυναμωθεί ούτε από το Brexit, ούτε πρέπει να αποδυναμωθεί με μείωση κονδυλίων για μεγάλα και φιλόδοξα σχέδια. Είναι σημαντικό να γίνει σωστός δημοσιονομικός σχεδιασμός ε, για να αποφευχθούν ε, τα υπερβολικά δάνεια και η υπερχρέωση που παρατηρήθηκε. Ε, Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό για να μην περιορίσουμε την ανάπτυξη ή να την καταργήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν κατάλληλες λύσεις ε, πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Η διαδικασία για την ε, θέσπιση του νέου πλαισίου πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν για να αρχίσουμε να συζητούμε για το επόμενο μέχρι το 2020. Πρέπει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Επίσης, ε, μια σταθερότητα των κανόνων είναι απαραίτητη για να είναι πιο αποτελεσματική η χρηματοδότηση. Η συνέχιση των κανόνων θα επιτρέψει αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα η Κομισιόν, στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, να τροποποιήσει όπου χρειάζονται τους κανόνες, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια κι εγώ στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τον κατάλογο των βασικών σημείων που αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγισή σας. Πιστεύω πραγματικά ότι αν υπάρχουν λιγότερα χρήματα για την επόμενη περίοδο, τι θα πρέπει να αναμένουμε. Ίσως θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ίσπραξης ε, ε, κονδυλίων ε, από τους ιδίους πόρους. Κατά πάσα πιθανότητα όμως θα υπάρχουν λιγότερα κονδύλια για την αναδιανομή στις διάφορες πολιτικές. Αν έχουμε λιγότερα χρήματα λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε στις μεγάλες προτεραιότητες της Ένωσης. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε την ε, γραμμή ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συμβολή στην ε, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και αποτελεσματικότητα των πόρων παράλληλα με την ευελιξία του μελλοντικού προϋπολογισμού και του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που είναι πιθανό να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Κάποιες ήδη ε, είναι, μπροστά μας. Πρέπει να προβλέψουμε χρήματα για τη μετανάστευση, την προσφυγική κρίση, την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Όμως πιστεύω ότι κάποιες από αυτές τις προσεγγίσεις μπορεί να συμπεριληφθούν στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Γιατί όλη η εμπειρία από την πολιτική συνοχής δείχνει ότι πρόκειται για μια από τις πολιτικές που μπορεί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν έχουμε ε, αρκετά ευέλικτη πολιτική συνοχής και πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και θα συνεχίσουμε να έχουμε επιτυχείς πολιτικές. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μπορεί να αναφέρομαι και την σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και Πολιτικής Συνοχής, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συστάσεις για κάθε χώρα που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, και έχουμε επίσης και την ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητα ε, και κάποια σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών και την υποστήριξη από την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, για την απλούστευση και την ευελιξία. Θα προσθέσω κάτι και για τις συνέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία και συνέργειες μεταξύ αυτής της πολιτικής και των άλλων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου περί των διαρθρωτικών ταμείων, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν θα πρέπει να χάσουμε από το, τη στόχευσή μας την πολιτική συνοχή, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και δημιουργικοί για να ε, δεχτούμε τη μελλοντική εξέλιξη αυτών των μέσων. Και βέβαια ε, και η διάρκεια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει η διάρκεια του Ίσως ε, θα πρέπει να δεχτούμε τη φόρμουλα των τύπο 5 συν 5 για να έχουμε μια επιλογή αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου ε, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις της Ένωσης. Σας υποστηρίζω λοιπόν και νομίζω ότι πράγματι πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Η κυρία Ανταμάτο η επόμενη σκιώδης, έχετε το λόγο. Πράγματι η έκθεση του συναδέλφου είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα όντας Βρετανός μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και το δύσκολο σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Ελπίζουμε να βρεθούν κάποιες λύσεις στα προβλήματα οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από ε, λογική και σεβασμό στα συμφέροντα των πολιτών και των δύο χωρών. Πάντως δεν θα πρέπει το πρώτο θύμα του Brexit να είναι η πολιτική συνοχής. Δεν θα πρέπει η πολιτική μας στον τομέα αυτό να μειωθεί ποσοστιαία λόγω της αποχώρησης και δεν θα πρέπει επίσης να αναμειχθεί με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την συνοχή η συμμαχία για τη συνοχή την οποία προωθεί η Επίτροπος και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνη. Ε, η Ρέτζη λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσει να πιέσει την έκθεση αυτή, να περάσει στην Ολομέλεια έστω και με δύσκολο τρόπο να υπάρξει αναφορά στον αποκλεισμό από εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει και από την Ολομέλεια. Ζητώ από τους συναδέλφους να είναι περισσότερο θαραλέοι, να κάνουν και άλλα βήματα, όπως το ζητούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να κάνουμε κριτική στους στόχους όταν δεν είναι οι σωστοί ε, να καταδικάσουμε τους νέους παράλογους, τις νέες παράλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά ταυτόχρονα να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Ένωσης. Η πολιτική συνοχή είναι βασικό μέσο χρηματοδότησης. ας μην την καταστήσουμε θυγατρική του σχεδίου Juncker. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική, πιο αξιοπιστή εξυπηρετώντας τα εδάφη και ελέγχοντας σωστά τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την πρόταση του συναδέλφου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Σας ευχαριστώ. Κύριε Όμερτζη, έχετε το λόγο. Θα ομιλήσω ως σκιώδης της ΓΚΟΕΝ. να ευχαριστήσω τον Βον για την παρουσίασή του. Πολλά είναι τα σημεία πάνω στα οποία συμφωνούμε και κάποια άλλα πάνω στα οποία έχουμε διαφωνίες. Πρώτον, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η πολιτική συνοχής επίσης, ε, ιδιαίτερα μετά το 2020, στα πλαίσια του Brexit toujours sur la raison pour laquelle la politique de cohésion γιατί η πολιτική συνοχής και ίσως και όλες οι πολιτικές της Ένωσης είναι αυτή που υφίσταται τι περισσότερες επιθέσεις και μάλιστα με τον πιο άδικο τρόπο. Ενώ είναι η πολιτική η οποία έχει πραγματικά μετριάσει στις περιφέρειες τις ε, επιπτώσεις της καταστροφικές της κρίσης του 2008 από πάρα πολλές άλλες πολιτικές οι οποίες καταστρέφουν δυστυχώς ε, τους θετικούς παραγωγικούς και εργασιακούς τομείς. Η πολιτική συνοχής λοιπόν είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζει τις αρνητικές συνέπειες που δημιουργούν οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών σαν παράδειγμα. Γιατί υφίστανται λοιπόν τέτοιου είδους επιθέσεις είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει αυτό το οποίο είναι η ουσία της, δηλαδή μια μεγάλη πολιτική αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια πολιτική. Η πολιτική συνοχής είναι η πολιτική αλληλεγγύης. Και αυτό ακριβώς έλεγε και η συνάδελφος Νταμάτο, παραμορφώνοντας την φύση της πολιτικής αυτής, πολλαπλασιάζοντας τα νέα χρωματοδοτικά μέσα από τη μία και από την άλλη, καθιστώντας την πολιτική συνοχής, θα έλεγα το θύμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των συστάσεων αναχώρα, στο τέλος φοβάμαι ότι δεν θα μείνουν και πάρα πολλά πράγματα. Συνεπώς θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις πρακτικές που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα, να συνεχίσουμε να αντιτιθέμεθα στις ε, ε, μακροοικονομικές αιρεσιμότητες όπως κάναμε μέχρι τώρα, γιατί αυτές πραγματικά θέλουν να υπονομεύσουν την πολιτική συνοχής. Πήραμε λίγο θάρρος, όχι και πάρα πολύ βέβαια, κατά τη διάρκεια του διαφθρωτικού διαλόγου Ας έχουμε όμως και το θάρρος να συνεχίσουμε την προσπάθεια επιβεβαίωσης των θέσεών μας, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε την καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση για το μελλοντικό πλαίσιο μετά το 2020, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε άλλη λύση από το να παραπέμπουμε στις αντιφάσεις τους μεν και τους δε. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο συμβουλίου. Θα πρέπει να δούμε ε, προς τα πού θα κλείνει η ζυγαριά. Θα επικρατήσει η λογική, δηλαδή η συνοχή, ή μήπως μέσα σε αυτή την ανοιχτή κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της ε, ε, προσπάθειας ε, επαναπροσδιορισμού των πολιτικών και μετά από αυτά που συνέβησαν και μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα σε πολλές χώρες, θα περάσουμε σε μια μεγαλύτερη περιφερικοποίηση των πολιτικών ή σε μια αμφισβήτηση των βασικών πολιτικών οι οποίες χαρακτηρίζουν την κοινή αγροτική πολιτική, την περιφερειακή, την πολιτική συνοχής, μεγάλα κομμάτια του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θα το δεχτούμε, αυτό θα επιτρέψουμε την πανεθνικοποίηση. Εμείς είμαστε οι Ρέτζοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μάχη. Εμείς είμαστε οι Ρέτζοι, πρέπει να δείξουμε θάρρος, να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας, να ψηφίσουμε με θάρρος την Ολομέλεια ήδη από την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει. Εδώ και καιρό κάνουμε κριτική στην πολιτική συνοχή με υπερβολικό τρόπο και παρόλα αυτά την χρησιμοποιούμε και ζητάμε την προστασία της για να πετύχουμε νέους στόχους, νέες προκλήσεις και πολλές φορές και νέες κρίσεις. Και πραγματικά αν δεν παρέμβει μέσω της πολιτικής συνοχής η Ένωση, κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει, ακόμα και για τη μεταναστευτική ε, κρίση, στην πολιτική συνοχή στα ρίξανε για να καλύψουν τις τρύπες. Πρέπει λοιπόν η πολιτική συνοχής να επιτρέψει να γίνουν οι διαφθορτικές αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν, αλλά όχι αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν αρνητικές καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη μάχη και πρέπει η πολιτική συνοχής να παραμείνει μια πολιτική αλληλεγγύης. Είμαστε έτοιμοι και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να σας πείσουμε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα του ε, χρηματοδοτικού πλαισίου. Νομίζω ότι στην σημασία της ε, πολιτικής αυτής ήδη υιοθετήσαμε μια έκθεση το θέμα είναι να διευκρινίσουμε το ποιες είναι οι θέσεις μας για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα εδώ να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η πρόταση την οποία κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στο λεγόμενο 5 5 και να καταστήσουμε μικρότερη και πιο μακριά, μακρά ταυτόχρονα την προγραμματική περίοδο, επιτρέποντας να υπάρξουν ευελιξίες εκεί όπου οι χρονισμοί το απαιτούν. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει ένα στατιστικό πλαίσιο για τις αλλαγές της πολιτικής συνοχής μετά την έξοδο των Βρετανών. Γιατί σαφώς και θα μειωθούν τα έσοδα, θα μειωθούν και τα έξοδα, γιατί και η Μεγάλη Βρετανία έπαιρνε πιστώσεις τέτοιου τύπου. Και ταυτόχρονα ε, θα αλλάξει και ε, ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών εισοδημάτων και θα αλλάξουν οι επιδοτήσεις προς διάφορες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο των αναγκών της πολιτικής συνοχής στο σύνολο της Ευρώπης μετά Brexit. Φυσικά στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να δούμε ε, ότι οι συμφωνίες με την ε, Ηνωμένο Βασίλειο να λαμβάνουν υπόψη ε, κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές οι οποίες θα μετακυλιστούν ίσως στην περίοδο μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, εξυπηρετώντας υποχρεώσεις που έχουν ε, αναλυφθεί στο παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι αν πράγματι θέλουμε να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχή στο εσωτερικό ενός προϋπολογισμού, ο οποίος θα έχει ανάγκη περισσότερους πόρους για να πετύχει νέους στόχους, που όλο ένα εμφανίζονται για την ανάπτυξη σαν παράδειγμα κοινή αμυντική πολιτική και σε άλλες πολιτικές οι οποίες ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες ε, ε, βρήκαν πόρους μεν αλλά δυστυχώς ανεπαρκείς ή πόρους οι οποίοι αφαιρούνται από τις υπόλοιπες χρηματοδοτούμενες πολιτικές μεταξύ των οποίων και κυρίως από τη συνεχή. Νομίζω επίσης ότι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε κυρίως είναι αυτό το οποίο θέτει το θέμα των ιδίων πόρων. Το θέμα των ιδίων πόρων θα πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα να βρούμε πόρους που δεν βαρύνουν άμεσα τον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά να βρούμε πόρους οι οποίες από τη μία πλευρά μας βοηθούν να πετύχουμε τους στόχους της COP21 σαν παράδειγμα, από την άλλη χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις λεγόμενες συνθήκες της εξωτερικής αγοράς οι οποίες πάρα πολύ συχνά αντιπροσωπεύουν θα έλεγα συμπεριφορές από ορισμένε χώρες ε, απαράδεκτες που απλά επιδοτούν οι χώρες αυτές τις βιομηχανίες τους και τα συμφέροντά τους. Και μάλιστα υπάρχουν και ε, φορολογικά συστήματα που επηρεάζουν την κατάσταση αυτή όπως ε, ο φόρος για τις ε, χρηματιστηριακές συναλλαγές, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο τον πολίτη αλλά την Ένωση να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι πόροι για τις νέες πολιτικές θα πρέπει να ευρεθούν κυρίως μέσα από τους ιδίους πόρους και όχι μέσω της αφαίρεσης πόρων από άλλες πολιτικές θεμελιώδεις για περιοχές ολόκληρες τις οποίες πολυθύμησαν και δεν θα επαναλάβω για λόγους χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να υπερασπιστούμε τη συνοχή, να πούμε ότι πράγματι απαιτούνται περισσότεροι πόροι, αλλά οι πόροι αυτοί θα πρέπει να ευρεθούν κυρίως μέσω του συστήματος των ιδίων πόρων, και όχι μέσω της ε, μεταφοράς της εσωτερικής ε, των πιστώσεων στο εσωτερικό του ιδίου του προϋπολογισμού. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αυτό με σαφή τρόπο προς τον συνάδελφο. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τον πόλεμο των φτωχών να τσακωνόμαστε για το ποιος θα δώσει τα χρήματα από τη μία πολιτική στην άλλη. Και εκεί θα έχει προβλήματα και η κοινή αγροτική πολιτική. Πάντως η κατάσταση αυτή που δημιουργείται λειτουργεί εις βάρος και της ΚΑΠ και της συνοχής για να εξασφαλίσουμε τις νέες δαπάνες. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο τους ιδίους πόρους έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε την άμεση φορολογική ε, θα έλεγα συνεισφορά των πολιτών και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους προστασίας παρόλα αυτά των βασικών αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών και να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις πολιτικές που έχουμε συμφωνήσει στο παρελθόν όπως έλεγχος της κίνησης των κεφαλαίων, ε, ρύθμιση των συνεπειών και μετρίαση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών, προβλήματα σχετικά με το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό dumping, θέματα τα οποία δυστυχώς δημιουργούν κάποιες χώρες εκτός της Ένωσης. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα συμφωνήσουν μαζί μας και θα πρέπει τα κράτη-μέλη επίσης να συμφωνήσουν και να υπερασπιστούμε έτσι λοιπόν την συνοχή μέσω κάποιων πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με έβρεση νέων πόρων. Γιατί αλλιώς ο κίνδυνος θα είναι να μειωθεί η πολιτική συνοχής. Μια πολιτική και θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα επί της ουσίας, μια πολιτική επαναλαμβάνω η οποία θα πρέπει σίγουρα σε κάποιους τομείς να ανασχεδιαστεί μετά την κρίση των τελευταίων ετών, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλειφθεί. Μια πολιτική που να συνδέεται καλύτερα με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, Μία πολιτική η οποία να συνδέεται καλύτερα με τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία πολιτική η οποία να βασίζεται στους ιδίους πόρους. Αλλά για να υπάρξει ένα απαιτούνται νέοι πόροι. Αν δεν υπάρξουν νέοι πόροι, τότε θα μείνουμε στα ίδια διαθέσιμα κονδύλια και αυτό είναι κάτι που δεν θα βοηθήσει τις λιγότερο φτωχές χώρες ε, δεν θα υπάρξουν ας πούμε πόροι για την ανταγωνιστικότητα που έχουν βοηθήσει πολύ τις λιγότερο ε, αναπτυγμένες περιφέρειες και δυστυχώς θα έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω και δεν θα επιτρέψουμε στις περιφέρειες αυτές να πάρουν μέρος στις κοινέ προσπάθειες. Θα έλεγα λοιπόν ότι στην φάση αυτή θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με όλα τα θέματα αυτά Τίθεται το θέμα επίσης και του προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Είναι κάτι το οποίο δεν άπτεται άμεσα της Επιτροπής μας, αλλά γνωρίζουμε ότι η πρόταση για ένα προϋπολογισμό της Ευρωζώνης είναι κάτι το οποίο μπορεί να θίξει ακόμα περισσότερο τη σύνοχη. Εφόσον λοιπόν υπάρξει ένας τέτοιος προϋπολογισμός και εγώ είμαι υπέρ, θα πρέπει όμως να βασίζεται σε μια προσθετική λογική και όχι σε μια ανταγωνιστική λογική με τα διαθέσιμα κονδύλια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια σχόλια κι εγώ. Εμπιστεύομαι ότι ο Ντέρεκ θα ηγηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην εμπειρία του και από τις συζητήσεις εδώ στο σώμα. Τώρα συζητώ πάρα πολύ με τις περιφέρειες στη χώρα μου. Και το κύριο μήνυμα που φτάνει από τις περιφέρειες τώρα είναι ότι θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα. Οπότε ας βρούμε έναν πιο έξυπνο τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Προς τη Σουηδική κυβέρνηση, για παράδειγμα, να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε. Θα μπορούσε να είναι και η δικιά μας προσέγγιση, λοιπόν. Γιατί με το που φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, που συνεισφέρει 10%, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άλλες χώρες πρέπει να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Συνεπώς, να το καταλάβουμε αυτό. Θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα, οπότε ας λειτουργήσουμε διαφορετικά. Με ένα πιο έξυπνο τρόπο, είτε πρόκειται για την έξυπνη δίκευση, είτε κάτι άλλο. Και να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορες ε, γενικές της διευθύνσεις να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους. χρησιμοποιούμε χρήματα από εθνικές ε, βέβαια πηγές από τις διάφορες χώρες, αλλά και από τα διάφορα ταμεία, τα ευρωπαϊκά, κοινωνικό, αναπτυξιακό, ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικής Ανάπτυξης και από εκεί δηλαδή μπορούν να υπάρχουν χρήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να στηρίξει πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Να δουλέψουμε δηλαδή πιο έξυπνα με λιγότερα χρήματα. Αυτή είναι η κύρια προσέγγιση μου εμένα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ποιος άλλος, η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για τις πολιτισμο οικονομικες προοπτικές μετά το 2020, υπάρχουν διάφορα ζητήματα για το μέγεθος, για τις προτεραιότητες, για τις αναλογίες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Και δεν ξέρω αν αυτές οι αβεβαιότητες κάποια στιγμή θα γίνουν βεβαιότητες. Στα πλαίσια του Brexit δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Κάποιοι συνάδελφοι στην Επιτροπή Προπολογισμών είπαν ότι ίσως χρειάζεται παράταση για δύο χρόνια αυτών των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Πολλά συζητιώνται δηλαδή. Και δεν είναι καλό για την πολιτική συνοχής. Ο χρόνος δεν ε, είναι υπέρ μας όσο περνάει. Το είπε και ο Λάμπερτ ότι πρέπει να πάρουμε σύντομα κάποια απόφαση για την επόμενη πολιτική συνοχής. Γι' αυτό και χαίρομαι που έχουμε θέσει τα βασικά και έτσι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει ήδη. Και τώρα πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες μέλη ώστε να δούμε ποια τελικά είναι ακριβώς η δικιά μας η θέση στα πλαίσια του, της νέας περίοδου. Ποιες είναι οι αβεβαιότητες, ποια είναι η θέση μας για την πολιτική συνοχής και όταν μιλάμε για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και την συνοχή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την νέα μας στρατηγική για το 2030. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και πώς εδέονται αυτές με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και την πολιτική συνοχή. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να περιμένουμε να έχουμε την πολιτική συνοχή μετά την απόφαση για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές εξαιτίας του Brexit. Και εξαιτία όλη αυτή τη αμφισβήτηση των σημερινών ε, πολιτικών δεν μπορούμε να περιμένουμε. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να φροντίσουμε να ακουστεί η φωνή μας, να αγωνιστούμε υπέρ της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε ποιες είναι οι ανάγκες. Η κατάρτιση, οι συνέργειες με άλλα μέσα, με άλλα εργαλεία, να αποφασίσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις επιχορηγήσεις ή άλλα ε, οικονομικά μέσα χρηματοδότησης και να ετοιμάσουμε το πλαίσιο για την πολιτική συνοχής έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι με τα διάφορα έγγραφα στατική σημασία, τα προγράμματα, ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να περάσουμε στην υλοποίηση. Αλλιώς εμείς θα φταίμε. Διότι θα διαχειριζόμαστε μία πολιτική η οποία δεν θα αποφέρει καρπούς. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλει κανένα άλλο το λόγο, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριε Γκίλεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Από πλούρας Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν, καλώς ορίζω την ε, συζήτηση. Ο κύριος Βόγαν έθεσε ε, διάφορα ζητήματα, όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στα περισσότερα από αυτά τώρα, δεν σας εκπλήσει αυτό. Τι να πω λοιπόν. Θα αρχίσω με το εξής. Βρισκόμαστε σε περίοδο προβληματισμού για το μέλλον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Υπάρχουν ε, διάφορα έγγραφα προβληματισμού που ετοιμάζονται και ένα σημαντικό για σας θα είναι εκείνο για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπη Κρέτου και την συνεργάζονται γι' αυτό και το περιμένουμε 28 Ιουνίου. ο κύριος Γιούγκερ, στην κατάσταση πραγμάτων για την Ένωση θα αναφέρει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πρόθεση είναι το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμπεράσματα στα τέλη της χρονιάς, να προσφέρει δηλαδή ένα πλαίσιο για αυτή την περίοδο προβληματισμού. Όσον αφορά τώρα ειδικά την πολιτική συνοχή, επιτρέψτε μου να πω και εδώ δύο λόγια και να απαντήσω. Στις συζητήσεις αυτές πάντα μιλάμε για απλοποίηση. Για να τα πω όσο πιο ανοιχτά μπορώ, πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί με το θέμα της απλοποίησης. Χρειαζόμαστε πιο σύντομες ρυθμίσεις και κανονισμούς και πιο ξεκάθαρους. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει και περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα αποτελέσματα. Παράδειγμα, υπάρχει μια παράγραφος στους κανονισμούς τώρα που ε, καθορίζει ποια είναι τα έγγραφα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Υπάρχει επίσης μια παράγραφος που μιλάει για την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό, όλοι ξέρουμε ποια είναι. Και αυτό που είπε ο κύριο Φανίστερο είναι αλήθεια, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή να κοιτάξουμε αποφασιστικά τους περιορισμούς που υπάρχουν και εμποδίζουν τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών και μεταξύ προγραμμάτων πιο πολύ μιλάμε με αυτούς που διαχειρίζονται τα προγράμματα, ακούμε ότι οι σημερινές ρυθμίσεις εμποδίζουν τέτοιες συνεργασίες, δεν τις ενθαρρύνουν. Συνεπώς όντως χρειαζόμαστε ένα πιο απλό πλαίσιο, πιο σύντομο, άρα θα είναι και πιο εύκολο να διαπραγματευτούμε πάνω σε αυτό. Αλλά βέβαια από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πιο μεγάλες ευθύνες οι χώρες μέλη, τα διαχειριστικά σώματα, γιατί ωραία δεν θα καθίσουμε να τα γράψουμε όλα στο χαρτί, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι χώρες θα έχουν την ευθύνη της απόδοσης των αποτελεσμάτων. Δεν θα υπάρχουν πάντα σαφείς απαντήσεις για όλα, άρα θα είναι δικιά τους ευθύνη. Αυτό το βήμα όμως πρέπει να γίνει και γρήγορα. Η κυρία Μάλετης νομίζω το στο τέλος ότι δεν είναι δυνατόν την επόμενη φορά να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση. 3-4% έχουμε δαπανίσει και είμαστε στα μέσα της περίοδου. Αλλά έτσι γίνεται κάθε φορά. Ε, δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να σταματήσει και νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο να αναλλάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάτι ήταν αυτό. Κάποια πράγματα μας τα είπατε. Εμείς αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η Κομισιόν εργάζεται και προετοιμάζει ένα κείμενο προβληματισμού τουλάχιστον. Το πρώτο το περιμένουμε τέλος Ιουνίου, σωστά, και θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Και ο κύριος Βον θέλει να ε, κλείσει τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ καλή συζήτηση. Κράτησα κάποια σημαντικά στοιχεία και καινούρια, τα κατέγραψα. Είναι πολλά, δεν θα τα αναφέρω όλα. Περιορίζομαι σε λίγα. Ο Λάμπερτ είπε ένα σωστό πράγμα, δηλαδή οι δυνατόν πρέπει να συμφωνήσω με το ταχύτερο δυνατόν για το ΠΔΠ, γιατί αυτό θα επηρεάσει τους κανονισμούς για την πολιτική συνοχή και όταν αρχίζει καινούριο πρόγραμμα πάντα υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή του και αν επιταχύνουμε τη διαδικασία λιγάκι αυτό θα ωφελήσει πάρα πολύ τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Οι συνάδελφοι συμφωνούν επίσης σχετικά στο 5 συν 5 Μερικοί βέβαια διαφώνησαν. Επίσης συμφωνούν για τους ίδιους πόρους. Όσοι μίλησαν για τους ίδιους πόρους είναι υπέρ. Για την απλούστευση συμφωνούν πολλοί, όπως ακούσαμε και από την Κομισιόν ε, και εκείνη αναγνωρίζει την ανάγκη ε, αυτή τη φορά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα απλουστεύσουμε τα πράγματα για όλους, για τους δικαιούχους, τις διαχειριστικές αρχές. Όλοι πρέπει να δουν τα αποτελέσματα της απλούστευσης αυτή τη φορά. Είναι σημαντικό για να φροντίσουμε η πολιτική συνοχής να γίνεται αποδεκτή στο μέλλον ως πολιτική σημαντική. Για τον προϋπολογισμό τον ίδιο, ε, μιλήσαμε για το μεγεθός του. Θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα σύστημα ιδίων πόρων. Η πολιτική συνοχή είναι κομμάτι του προϋπολογισμού. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να δείξουμε την επιτυχία της πολιτικής συνοχής και όπως είπες και εσύ Λάμπερ να δείξουμε ότι η πολιτική συνοχής βοηθάει την Ένωση να επιτύχει και άλλους στόχους και μας πάει στο επόμενο θέμα αυτό, τις συνέργειες να με κονδύλια της πολιτικής συνοχής με άλλα, είτε είναι Horizon 2020 είτε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για να ε, έχουν αντίκτυπο όλα τα κονδύλια, αλλά να επιτυγχάνουν και τους στόχους της Ένωσης. Αυτά είναι κάποια σημεία που ήθελα να αναδείξω, υπάρχουν και πολλά άλλα μου φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλη η έκθεση αυτή. Θα συμπεριλάβω τις απόψεις των συναδέλφων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα έχω ένα κείμενο ε, τον Ιούνιο την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε το σχέδιο της γνωμοδότησής σας ε, για την συνάντηση του Ιουνίου. Οπότε τελειώνουμε τη συζήτηση αυτή και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι οι ε, εδαφικές τυπολογίες, τέρκετ. Πρόκειται για τον κανονισμό ΝΑΤΣ εδώ. Ο τωρινός κανονισμός ΝΑΤΣ δεν καλύπτει τις εδαφικές τυπολογίες ως ε, ορισμούς ε, αστικών, ε, αγροτικών, παράκτιων και άλλων περιοχών. Είναι καινούργιε οι τυπολογίες, παρόλο που τις χρησιμοποιούμε στις συζητήσεις. Το θέμα το θέτουν οι προτάσεις της Κομισιόν για τις τυπολογίες και η πρώτη συζήτηση για το θέμα έγινε στη συνάντησή μας του Απριλίου. Τότε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μας εξήγησε το πώς έχει το θέμα και τι σκοπούς εξυπηρετεί η πρόταση. Η αρχική μας θέση ήταν ότι ήταν μια ε, εύκολη τεχνική πρόταση που θέλαμε να εγκρίνουμε χωρίς τροπολογία με απλουστευμένη διαδικασία. Αλλά Τώρα συζητούμε για δεύτερη φορά το θέμα αυτό και αυτό γίνεται επειδή το Συμβούλιο τώρα ε, ε, πήρε θέση σε επίπεδο ομάδας εργασίας και κατέληξε ότι η πρόταση θα χρειάζεται τροποποίησης. Οι βασικές αλλαγές είναι η υποχρέωση υποβολής έκθεση από την Κομισιόν και το διάστημα στο οποίο πρέπει να υποβάλλεται και επίσης φαίνεται το Συμβούλιο να ισχυρίζεται ότι για στατιστικούς λόγους η Κομισιόν δεν μπορεί να αλλάζει τις, τον κατάλογο των περιφερειών εκτός και αν τα κράτη-μέλη τα οικία κράτη-μέλη έχουν ε, ενημερώσει για τις σχετικές αλλαγές την Κομισιόν. Δύο τρόπο έκανε λοιπόν η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Αντιλαμβανόμεθα ότι η Κομισιόν ε, έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις και αυτό την καλέσαμε να έρθει, να εξηγήσει τις θέσεις της και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση. Πρώτα θα πάρουν το λόγο οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και μετά θα πάρουν το λόγο οι σκιώδες για να κάνουν ερωτήσεις εάν είναι εδώ. Και μετά θα αποφασίσουμε τι συνέχεια θα δοθεί, αν δηλαδή θα επιμείνουμε στη θέση μας ενάντια στις αλλαγές και βραχύτερη διαδικασία και αν θα προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο με αυτή τη θέση ή αν μπορούμε να τροποποιήσουμε την πρόταση. Δίνω το λόγο στον κύριο Σέφερ. Εσείς θα αρχίσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε το θέμα το συζητήσαμε πολύ στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Και τρεις μεγάλες αλλαγές υπάρχουν. Η πρώτη που δεν την αναφέρατε, συγγνώμη που συμπληρώνω εδώ, η πρώτη λοιπόν είναι να μην επηρεάσω με κανένα τομέα πολιτικής, αφού αυτή είναι μια στατιστικής φύσεως πρωτοβουλία και στην αρχική πρόταση είχαμε πει ότι θέλουμε να διευκολύνουμε τις ε, αποφάσεις ε, και τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Συμφωνήσαμε να βγει αυτό γιατί δεν έχουμε πρόθεση να παραβλάψουμε κατ' ουδένα τρόπο οι ασδήποτε πολιτικές αποφάσεις με την πρωτοβουλία μας αυτή. Το δεύτερο θέμα είναι ότι από την πλευρά της Κομισιόν δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό το δεύτερο γιατί αφορά τις αλλαγές και πάντοτε λειτουργούμε βάσει πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και συζητούμε με τα κράτη-μέλη αυτές τις αλλαγές και αυτό γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο τώρα στην πρόταση του Συμβουλίου, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου εννοώ πάντα. Και πρέπει να πω ότι δεν έχουμε καμιά απολύτως δυσκολία ή επιφύλαξη με την πρόταση αυτή η οποία ε, υπάρχει στην πρόταση του Συμβουλίου που έχετε μπροστά σας. Το, το τρίτο θέμα αφορά την πενταετή διάρκεια από πλευράς κομισιών Έχουμε μάλλον ουδέτερη θέση, γιατί το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει τη θέση, θα πάρει. Το Συμβούλιο μίλησε για τον περιορισμό των πέντε ετών με την έκθεση και την συνέχιση μετά την έγκριση. Η Κομισιόν είχε προτείνει απεριόριστο χρονικό διάστημα και θα ήθελε να αφήσει το θέμα στα χέρια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση που αρχίζουμε. Ελπίζαμε να πάει ομαλά, αλλά οι σκιώδεις οι συγητές, οι όσοι τέλος πάντων βρίσκονται εδώ, αν έχουν να πούνε κάτι, έχει καλώς, αλλιώς θα οργανώσω συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές για να καθορίσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Ίσως αυτός θα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Έτσι. Τίποτα άλλο τώρα. Όχι γι' αυτό. Καλώς, συνεπώς θα οργανώσω συνάντηση με τους σκιώδες εισηγητές από αυτού και θα αποφασίσουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με ό,τι προτάσεις έχουμε του Συμβουλίου, της Επιτροπής, θα την ακούσουμε και έτσι θα δούμε πώς θα καθοριστεί δικιά μας η θέση για τη στήριξη της πρότασης επιτροπής χωρίς τροπολογίες και να πάμε σε τριμερή διάλογο ή αν θα τροποποιήσουμε την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών τώρα. Είχαμε συνεδρίες των συντονιστών χτες το απόγευμα και έχετε πάρει με email τις αποφάσεις. Εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Ναι, καλώς. Ευχαριστώ. Διάφορα. Έχουμε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Καλώς. Υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου το απόγευμα και την επόμενη μέρα το πρωί στις 20. Αυτά. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, για τη βοηθειά τους. Κλείνω τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.